Πολλή δουλειά να κάνουμε. Και τώρα μερικά ενημερωτικά. Σας επισημαίνω ότι η κυρία Σακίνης Ασιάδη η οποία καταδικάστηκε εις θάνατο στο Ιράν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που λάβαμε, ε, πέτυχε την ακύρωση της απόφασης από το ανώτατο δικαστήριο. Υπέστη μαστίγωση 99 φορές, είπε στου 99 μαστιγώσεις και έγινε αυτή η προσφυγή στις Ελληνές Αρχές εκ μέρους της Ευρώπης τόσο ώστε να ακυρωθεί αυτή η ποινή και το, το κοινοβούλιο είναι κατά της ε, θανατικής ποινής ανεξαρτήτως κατηγορίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, τα πρακτικά της Συνόδου της 8ης Ιουλίου για τα οποία σας